Θέλω να ανακοινώσω το εξή ότι η Επιτροπή ΙΜΚΟ έχει καταθέσει μια σύσταση να μην υπάρξει αντίρρηση στις καταξισιοδότηση πράξεις. Αυτό ανακοινώθηκε χθε. Δεν υπήρξε καμία ε, αντίρρηση μέσα στο διάστημα των 24 ωρών που προβλέπεται. Βάσει του άρθρου 105.6 η σύσταση αυτή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα δημοσιευτεί αύριο με τα πρακτικά της αυριανής συνεδρίασης του Κοινοβουλίου. Βάσει της ημερησίας διάταξη. περνούμε τώρα στο